δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για τα, την ε, κατάσταση στη Λιβύη. Να δώσω το λόγο. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό, οπότε περιμένουμε για να έρθει. Κύριε Υπουργέ Κούντερς, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μαζί ένα σημαντικό θέμα από πλευρά τη υπάτηση εκπροσώπου Φεντερίκα Μογκερίνη. Είναι η κατάσταση στη Λιβύη. Τι πρόοδο έχει σημειωθεί και τι προκλήσει έχουμε ενώπιόν μας. Έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδο από την προηγούμενη φορά που το συζητήσαμε εδώ το θέμα. Έχουμε την ε, πολιτική συμφωνία που υπεγράφει στο ΣΚΙΡΑΤ στις 17 Δεκεμβρίου. Το Προεδρικό Συμβούλιο ε, ε, έχει συσταθεί και εργάζεται και η κυβέρνηση Εθνικής Συνένεσης και το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκαν μόλις μπόρεσε την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου η κυρία Μογκερίνη πήγε στην Τίνιδα να συναντήσει το Προεδρικό Συμβούλιο για να εκφράσει την πολιτική συμπαράσταση της Ένωσης και για να συζητήσει με όλα τα μέλη για τις άμεσες και μακροπρόθεσμες ενέργειες που μπορεί να κάνει η Ένωση για να στηρίξει τις λιβικές αρχές. Τους επιθυμήσαμε ότι έχουμε εδώ και καιρό έτοιμο ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και το μόνο που χρειάζεται είναι να αρχίσει να λειτουργεί εντός της χώρας η κυβέρνηση εθνικής συνένεσης. Διάφορες νέες ανακοχές υπεγράφησαν πρόσφατα μεταξύ διαφόρων δήμων, μεταξύ της Μισράτα και του Ταγουάργα που είναι κοντά, οπότε σταμάτησαν οι εχθρότητες και εχθροπραξίες που είχαν ξεκινήσει από την Επανάσταση του 11 μεταξύ Ζαβίγια και Ζιντάν, δυτικά της Τρίπολης, στο Σουρμάν, ε, δυτικά της Τρίπολης και στο Νότο. Ε, είναι ακόμη εύθραυστη η ανακοχή μεταξύ των Τούμπου και των Τουαρέκ που εδώ και μήνες ε, ήταν, είχαν εχθροπραξίες στο Τουμπάρι. Όμως ε, έστω και προσωρινά αναγνώρισαν ότι αυτή η διαδικασία από την αιγύδα των ΗΠΑ είναι η μόνη ερευνητική διαδικασία. Το σώμα των αντιπροσώπων δεν ενέκρινε τις υπουργικές, ε, τους υπουργικούς διορισμούς στην κυβέρνηση, στην προτινόμενη κυβέρνηση Εθνικής Συνένεσης. Χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις. Αλλά ελπίζουμε και αναμένουμε ότι τελικά οι υπεύθυνοι στη Λιβύη θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση. Πρέπει να υπάρχει μια ενωτική κυβέρνηση που να εκπροσωπεί όλε τι περιοχέ, όλε τι πολιτικέ ομάδε. Μόνο μια τέτοια κυβέρνηση μπορεί να δώσει πραγματική ελπίδα στου Λιβύου ότι η χώρα του θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια για πάντα την εξάπλωση τη τρομοκρατία, την οικονομία που είναι στα όρια τη αβίσου και την ανάγκη ανάπτυξη όταν θα εγκριθεί η κυβέρνηση εθνική Ενότητας από το Κοινοβούλιο, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ασφάλεια του πληθυσμού και η καταπολέμηση του ΝΤΑΕΣ. Η ασφάλεια πρέπει να ε, είναι αντικείμενο της ε, δράσης των ίδιων των Λιβύων. Αυτή θα είναι οι νέε δυνάμει ασφαλείας, ενώ η διεθνή κοινότητα μπορεί να δώσει περισσότερη βοήθεια και εκπαίδευση αν το ζητήσει η Εθνική Κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στι ε, προσπάθειε διασφάλιση τη ασφάλειας μέσω της ε, μονάδας μας στην Τίνιδα. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις προσπάθειες των ΗΠΑ και των ε, αρχών της Λιβύης. Και συμφωνήσαμε αυτός ο πυρήνας μας να ενισχυθεί και να βελτιώσουμε και τις δυνατότητε ε, πολιτικού σχεδιασμού μέσω της διεύρυνσης της αποστολής UBAM. Θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί τις επόμενες εβδομάδες και να δώσει Περισσότερε δυνατότητε για στήριξη τη αστυνομία και για την καταπολέμηση τη τρομοκρατίας, την ασφάλεια των συνόρων, τα τελωνία και την μετανάστευση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η δημοκρατική μετάβαση στη Λιβύη είναι δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Αλλά αυτή η συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκαν τα Ηνωμένα Έθνη έχει αποτελέσματα, πρέπει να συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε. Για την εναλλακτική λύση είναι απλά το χάος. Μια χώρα στα όρια της οικονομικής κατάρρευση. Όλα αυτά όμως μπορούμε να τα αποφύγουμε. Είναι καθήκον μας ως ε, γείτονε της Λιβύης να συνεχίσουμε να στηρίξουμε την διαδικασία των ΗΠΑ και το GNA, το Εθνικό Γενικό Συμβούλιο, έχει δεσμευτεί ότι θα στηρίξει αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Τώρα θα έπρεπε να δώσω το λόγο στον κύριο Μπροκ, αλλά δεν τον βλέπω. Α, θα μιλήσει η κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Σήμερα πράγματι η προτεραιότητα στη Λιβύη είναι ο σχηματισμός ε, κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης. Ε, και επίσης θα πρέπει να, να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες του Μαρτίν Κομπλέρ. Η διαδικασία στη Λιβύη είναι πάρα πολύ σημαντική για να δοθεί ένα τέλος ε, στην ε, ε, πολιτική διαίρεση και στο διχασμό που ισχύει και σε γεωγραφικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση στη Λιβύη και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και την ευθύνη των λιβικών κομμάτων και ενώπιον των Λιβύων αλλά και των άλλων χωρών του Σαχέλ συμπεριλαμβανομένες και της Μπουργκίνα Φάσο και του Μαλή. Του Μάλι. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό λοιπόν παράγοντα και σε περιφερειακό και σε διεθνέ επίπεδο και αυτή τη στιγμή είναι αποφασιστική σημασία να προχωρήσει η κατάσταση στη Λιβύη. Η βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνούς κοινότητα είναι να είμαστε έτοιμοι σε διάφορα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή συσταθεί κυβέρνηση ε, με ε, νέα αποστολή βοήθεια στα σύνορα ή ε, μια νέα πολιτική αποστολή η οποία θα πρέπει να αποσταλεί εκεί ταχύτατα. Θα πρέπει επίσης να κινητοποιήσουμε ήδη τη διεθνή κοινότητα για την οικονομική ανοικοδόμηση, διότι ε, εάν η οικονομία της χώρας ε, βυθιστεί, η κυβέρνηση θα είναι τελείως αδύναμη και ανίσχυρη. Επίσης, θα πρέπει να ε, υποστηρίξει η διεθνή κοινότητα οργανωμένα τη Λιβύη. Τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αφρικανική Ένωση, η Ένωση των Αραβικών Κρατών μπορούν όλοι να συνεισφέρουν για την ανοικοδόμηση και την πρόληψη τη ριζοσπαστικοποίηση, για παράδειγμα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ώστε η κατάσταση στη Λιβύη να μην επιδεινωθεί έτσι περαιτέρω για όλου μα. Ευχαριστώ, ο κύριο Μποστινάρου, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κούντερς, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι τελευταίες πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη Λιβύη δείχνουν μια χώρα στο χείλος της Αμπίσου. Το είπατε και εσείς προηγουμένω. Ε, κανείς δεν ξέρει σε για πολλωστή φορά, για πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Καταστροφική κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί. Το Ντάος έχει καταστρέψει τους δρόμους και είχε επιτόπου κάποιες εκατοντάδες μαχητές, τώρα όμως φαίνεται ότι έχει χιλιάδες. Είναι λοιπόν εύκολο να κατανοήσει κανείς ε, τι σημαίνει το να προσπαθήσει κανείς να τους εξαφανίσει. Η πολιτική λύση είναι απαραίτητο να βρεθεί επιτακτική και απευθυνόμαστε ε, στους, στο Κοινοβούλιο για να επιδείξει συμβαστική διάθεση και από τη στιγμή που θα προταθεί ο κατάλογος των Υπουργών, ελπίζουμε τι επόμενε μέρε, ώρε ώρες μάλλον, να γίνει αποδεκτό. Αυτό είναι ένα μικρό βήμα στη σωστή κατεύθυνση, διότι οι προκλήσει μπροστά μα είναι πάρα πολλέ. Ε, δεν θα ήθελα να ξεχάσω και κάτι άλλο σημαντικό. Μέχρι τώρα οι κυρώσεις έναντι κάποιων ανθρώπων εκτοξεύτηκαν αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Τώρα πια έχει έρθει η στιγμή να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να εφαρμόσουμε κυρώσεις έναντι εκείνων που υπονομεύουν την πολιτική λύση για τη Λιβύη. Η νέα κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει την ολέτρια ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα ε, για να γίνει αυτό χρειάζεται τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας. Σήμερα το πρωί ο κύριος Μπουχάρη, ο πρόεδρος της Νιγηρίας, είπε ότι η κατάσταση στη Λιβύη δεν είναι μόνο ένα τοπικό περιορισμένο πρόβλημα, καθίσταται σημαντικό περιφερειακό πρόβλημα με ουσιαστικές συνέπειες σε μια περιοχή η οποία ήδη έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Σήμερα λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει ενωμένο στρατός για να εξαφανίσει τον Ντάεσ, αλλά αν ε, δεν γίνει αυτό θα πρέπει να βοηθήσει και η διεθνής κοινότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ ο κύριος ε, Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε αισιόδοξοι ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε το Δεκέμβριο του περασμένου έτου θα εφαρμοστεί πλήρω και ότι θα υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση ε, που θα σχηματιστεί. Τέτοιου είδου συζητήσει βέβαια είναι χρονοβόρε και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αυξανόμενη παρουσία του ISIS στην περιοχή. Ε, στη Ρώμη συναντήθηκαν ε, οι σύμμαχοι και οι Λιβύη είναι θέμα που του απασχολεί. Όλε οι δυνατότητε πρέπει να παραμείνουν ανοιχτέ. Εγώ καλωσορίζω το γεγονό γεγονός ότι οι ΗΠΑ σκέπτεται να στείλει στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη όπως έγινε και στη Συρία. Ε, η έκθεση δείχνει ότι η γαλλική κυβέρνηση ε, δεν έχει αποκλείσει και άλλη στρατιωτική επέμβαση και ελπίζω και το Ηνωμένο τελικά και αυτό να σκεφτεί να στηρίξει τέτοιου είδους ενέργειες γιατί δραστηριοποιούμεθα ή δραστηριοποιηθήκαμε για να πέσει ο Γκαντάφη. Υπάρχουν κενά στις ακτές ε, της Λιβύης μετά την ήττα που υπέστη αυτή στη Συρία. Άρα δηλαδή είναι κίνδυνος ε, ασφάλειας για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τελίτσκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες για το σχέδιο ψηφίσματος που καταφέραμε να συζητήσουμε και επί του οποίου συμφωνήσαμε. Πρόκειται για ισορροπημένο κείμενο και υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από όλες τις πλευρές και ελπίζω να αποδειχθεί αυτό και αύριο κατά την ψηφοφορία. Ακούστηκε ήδη σήμερα ότι ο πρόεδρος Μπουχάρη μας υπενθύμησε ε, την κατάσταση όχι μόνο στην Νότια Λιβύη, αλλά και ε, το γεγονός ότι όλη η περιοχή του Σαχέλ βιώνει κρίση. Και επίσης να πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση όπλων από ό,τι ποτέ στην περιοχή. Επίσης ε, γίνεται διακίνηση ανθρώπων τον τελευταίο, τα τελευταία χρόνια και εντατικοποιείται. Υπάρχει πρόβλημα και για μειονότητες και για μετανάστες. Η κατάσταση είναι ολέθρια και τραγική. Πρέπει λοιπόν επιτέλους να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αλλά φυσικά ε, πρέπει να, να υποστηριχθεί η συμφωνία στη συνέχεια. Και τι πρέπει να κάνουμε για να υποστηρίξουμε και τη Λιβύη. Είναι προϋπόθεση εκ των όνου κάνευ ότι θα ε, πρέπει να επικοινωνούμε μόνο με όσους ε, προσπογράφουν τη συμφωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη, κάποιοι πολιτικοί βρίσκουν ανεπίσημους διάβλους για να συνεργαστούν και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Το Ισλαμικό κράτος είναι παρόν. Ένα τμήμα της ακτής είναι ουσιαστικά στα χέρια του Ισλαμικού κράτους και η περιοχή δεν απέχει πάρα πολύ από την Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις για μια ευρύτατη σύραξη στην οποία θα κερδίσει συνεχώ έδαφο το Ισλαμικό κράτο. Δεν πρέπει λοιπόν να επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος, πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν καλύτερα την κατάσταση σήμερα. Δεν θα είναι εύκολο, πρέπει όμως να υπάρξει υποστήριξη και για μένα η ίστατη λύση, αν ε, αποτύχουν οι πολιτικές προσπάθειες, θα είναι τελικά παρέμβαση. Ε, καταλαβαίνω ότι δεν έχουν κορυφωθεί ακόμα οι δράσεις κατά του Ισλαμικού κράτους, αλλά αυτή είναι η τελευταία μας ε, λύση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούσο Περμούη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες για την εφαρμογή της πολιτικής συμφωνίας στη Λιβύη ε, που επιθυμεί ο ΙΕ. Πρόκειται για κάτι το οποίο ε, σιγά σιγά οδηγεί κάποιους να θέλουν να εγκαταλείψουν αυτή την αργά γη αλλά ασφαλή οδό και να πάμε πλέον και πάλι και να ακούσουμε την πνοή του πολέμου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ε, είναι υπέρ μιας νέας στρατιωτικής παρέμβασης. Θα πρέπει να θυμηθούμε τι έγινε με την προηγούμενη στρατηγική παρέμβαση του ΝΑΤΟ που κατέστρεψε πλήρως ε, τη Λιβύη, χιλιάδες αθώα θύματα και πλήρης ε, αποσταθεροποίηση της περιοχής και επέκταση της τρομοκρατίας. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε στρατιωτική παρέμβαση, απορρίπτουμε την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και ζητάμε να σταματήσει οποιαδήποτε εξαγωγή όπλων και η χρηματοδότηση των παραστρατιωτικών ομάδων, δηλαδή να μην αγοράζουμε το πετρέλαιό τους και να ε, εφαρμοστεί το ψήφισμα 1970 ε, το Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η κυρία Λοχμπίλερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πιο επίγον καθήκον της Ένωσης είναι να βοηθήσει τα Ηνωμένα Έθνη για να υπάρξει μια ενιαία κυβέρνηση. Οι διάφορες ομάδες πρέπει να αποδείξουν ότι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να υπάρξει μια ενιαία κυβέρνηση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Είναι αναμφίβολο ότι στι διαπραγματεύσει ορισμένε ομάδε του πληθυσμού και πολιτοφυλακέ δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Αλλά α είμαστε ρεαλιστέ. Χωρί μια κοινή δράση των κυβερνήσεων στην Τρίπολη και το Τομπρούκ δεν θα υπάρξει ειρήνευση. Παρατηρούμε ότι στο χάος που επικρατεί στη Λιβύη το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Γι' αυτό πρέπει όλες μας οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στην καταπολέμησή του. Όποιος όμως νομίζει ότι μέσω στρατιωτικής ε, επέμβασης μπορεί να το, να το επιτύχουμε αυτό, κάνει λάθος. Λόγω της χαοτικής κατάστασης όχι μόνο θα αποτύχει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, στην ουσία θα είναι βούτυρο στο ψωμί εκείνων των ομάδων που θεωρούν ότι οποιαδήποτε διεθνής προσπάθεια είναι παραβίαση της ε, κυριαρχίας της χώρας και θα το αξιοποιήσουν προπαγανδιστικά και η λεγόμενη τρίτη φάση της παρέμβασης ε, των ε, Ηνωμένων Εθνών για να αντιμετωπιστούν οι διακινητές είναι αμφισβητήσιμη γιατί στην ουσία θα υποδαβλήσει την ε, περαιτέρω τη σύγκρουση. Ξέρουμε ότι πολλοί απάγονται, βασανίζονται και αυξάνεται η βία κατά των δημοσιογράφων και οι μετανάστες ζουν σε άθλιες συνθήκες. Δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε αυτό η διεθνής κοινότητα. Δεν θέλει να υπάρξει δεύτερη Συρία. Αν δεν το θέλουμε αυτό, πρέπει να βοηθήσουμε με ανθρωπιστική βοήθεια τη μελλοντική κυβέρνηση και τι ε, οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε οι υπεύθυνοι για σοβαρέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα λογοδοτήσουν σε διεθνή δικαστήρια. Ευχαριστώ. Υπάρχει μία. Ε, υπάρχει μία μπλε κάρτα. από τον κύριο Τάνοκ για τον κύριο Κόουσο, αλλά ε, με συγχωρείτε έχει περάσει τώρα δεν μπορούμε να την ε, να τη δεχθούμε με συγχωρείτε έχει περάσει σειρά σας ο κύριος Καστάλντο τρία λεπτά Πώς το καταφέρατε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική στις μέρες μας ε, πάσχει από το σύνδρομο του κάνω. Να κάνω οτιδήποτε προκειμένου να μην δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε ακίνητοι και να μας ξεπεράσει ο ανταγωνισμός ή τα γεγονότα. Ένα από τα χρόνια νοσήματα είναι αυτά τα οποία κάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας μου, ο κύριος Ματέο Ρέντσι. Υπάρχουν πολύ σοβαρά όμως ε, ε, αποτελέσματα. Όπως για παράδειγμα το να δώσουμε το πράσινο φως ε, για μια στρατιωτική παρέμβαση ε, και αυτό είναι ασυγχώρατο για επικεφαλής μια χώρας. Και πραγματικά το να καταστρέψουμε μια χώρα είναι έγκλημα. Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε από το 2011 και τα όσα συνέβησαν στη συνέχεια ήταν άμεση συνέπεια των όσων έτρεσαν τόσο απερίσκεπτα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιέστηκε να κάνει την παρέμβαση. Την πίεσε η κυβέρνηση για να βάλουν τα χέρια τους ε, στο πετρέλαιο ε, από την Ιταλική Έννη, να αυξήσουν την παρουσία τους εκεί και τη στρατιωτική παρουσία και στο εσωτερικό και του ίδιου του Σαρκοζή και να προλάβουν το πιθανό σχέδιο του Καντάφη για να σταματήσει ε, το πρόγραμμα μεταξύ Γαλλίας και Αφρικής με μια παναφρικανική συνεργασία με βάση τα αποθέματα πετρελαίου της Λιβύης. Όλα αυτά έγιναν με υποκίνηση των ΗΠΑ. Οι παρεμβάσει τη Γαλλία, τη μεγάλη Βρετανία, τη Ιταλία και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έγιναν κατανοητά. Ε, πρόκειται για αρχηγούς κρατών που ε, προσπαθούν να δώσουν απαντήσει μετά τα γεγονότα στο Παρίσι, να δείξουν του μίστου ο ένας τον άλλον και φαίνεται ότι το Ισλαμικό κράτο κατάλαβε τώρα που το απείλησαν. Προσπαθούν να ε, προστατεύσουν τα πετρελαϊκά αποθέματα και όχι την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Και φυσικά στόχο είναι να μην χάσει κανεί τι εκλογέ. Προτεραιότητα είναι να σταθεροποιηθεί η Λιβύη, να ξαναξεκινήσει η διαδικασία μετάβαση. Εάν εμεί ξαναβορβαδίσουμε και αναπτύξουμε τα στρατεύματά μας, ουσιαστικά θα συμμαχίσουν τα, οι Ισλαμικές παραστρατιωτικέ ομάδες γύρω από το Ισλαμικό κράτος, Όπω έγινε μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ υπάρχει λογική της εκδίκησης αντί της συμφωλήσης και να πώς αυξάνεται το Ισλαμικό κράτος ε, με τους πρώην ε, συμμάχους του Καντάφη. Όλα αυτά από πολιτικά σφάλματα. Αν παρέμβουμε χωρίς σαφή πολιτική συμφωνία οι παραστρατητικέ ομάδες που θα αντιμετωπίσουν τις δικές μας δυνάμεις ε, θα θεωρηθούν ότι είναι κατά των ε, εισβολέων και ε, θα υποσκάψουν ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της συμφιλίωσης. Θα πρέπει οι περιφερειακές δυνάμεις ενώπιον αυτού του αυξανόμενου χάους να σταματήσουν πλέον να παρεμβαίνουν και να μην τους δελεάζει η λογική των ισχυρών που απλώς υποσκάπτουν τι διαπραγματεύσεις. Αν πραγματικά λοιπόν θέλουν να βοηθήσουν θα πρέπει να μιλήσουν με τις τοπικές ε, αρχές και με την πραγματικότητα εκεί. Να αποφύγουμε λοιπόν την καταστροφή και την κατεπίγουσα κατάσταση και πρέπει να δώσουμε ε, μία μάχη και να επιτύχουμε αυτό το οποίο είναι δίκαιο. Ο κύριος Μποργέτσιο για δύο λεπτά και δυόμιση λεπτά. Σήμερα λοιπόν έχουμε με τον Τομπρού μία επιστολή προς εμάς ε, και κρίμα που δεν είναι εδώ είπατε εκπρόσωπος. Εκεί λοιπόν το κοινοβούλιο του Τομπρού μας λέει ότι δεν είναι σε θέση λόγω του εμπάργου να ε, αμυνθεί έναντι του Ισλαμικού κράτους. Ε, υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις οι οποίες ενδιαφέρονται να ελέγχουν τους, τις πρώτες ύλες της Λιβύης. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή δεν να κάνει τίποτα για να βοηθήσει τη Λιβύη να αντιμετωπίσει το Ισλαμικό κράτος που έχει φτάσει και στις πόρτες της Ευρώπης ε, ε, η επέμβαση γαλλοαμερικανική ε, δεν ήταν αποτελεσματική. Μήπω λοιπόν πιστεύει, είπατε εκπρόσωπο ότι θα πρέπει να υπάρξει άλλη μία προσπάθεια γιατί αλλιώ οι Λίβοι θα χάσουν τελείω τον έλεγχο των συνόρων του και έτσι θα υπάρξει μία περαιτέρω απόβαση στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν το εμπάργκο, υπήρχε και τότε κατά του Καντάφη, αλλά έχει καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν υπάρχει πια ο Καντάφη. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εμεί λοιπόν ζητάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατη να υπογράψουν συζητούν τις συμφωνίες επανιστοχής όπως αυτό που έχει η Ιταλία με τη Λιβύη για τα Ηνωμένα Έθνη ε, 400.000 ε, πρόσφυγες είναι έτοιμοι να έρθουν στην Ευρώπη ε, και όπως είπε ο Γάλλος υπουργό, εκεί θα μπορούσαν να δυσδύσουν πάρα πολλοί τρομοκράτες ε, κάποιοι εν που έχουν σχέσεις με το Ισλαμικό κράτος. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η έκκληση που έρχεται από τους βουλευτές του Τόμπρου, του Κοινοβουλίου του Τόμπρου αυτή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το δικό μας το Κοινοβουλίο. Αυτή είναι η επιστολή και βεβαίως ε, θα ήθελα αυτή την επιστολή να την παραδώσω στην ε, είπατε εκπρόσωπο που μέχρι τώρα κόφευσε σε αυτές τις εκκλήσεις. Dodge για δύο λεπτά. Ένα λεπτό. Στην δική μου την περιφέρεια, στην Βόρεια Ιρλανδία και για όλα τα θύματα. Είχαμε πολλές φορές ε, εγκλήματα από τον IRA και προσπαθούμε ακόμη να αγωνιστούμε για να αποζημιωθούν τα θύματα. Και υπάρχουν επικρίσεις προς τον Πρωθυπουργό Τόνι Μπλέα, τον πρώην Πρωθυπουργό, που δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις σε σαφείς ερωτήσεις για τις συζητήσεις που έκανε για την αποζημίωση για τα θύματα του IRA όταν ο συνταγματάρχης Καντάφη ήταν ακόμη στην εξουσία. Διότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι νόμες ανησυχίες των θυμάτων της τρομοκρατίας. Πρέπει σίγουρα να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη για να μπορέσουμε να έχουμε ε, σωστές αποζημιώσεις από τη Λιβύη για τα θύματα αυτά. Θέλουμε μια ειρήνη. Θέλουμε να υπάρχουν θεμελιώδεις ελευθερίες. Θέλουμε να υπάρχει περιθώριο για να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους οι θρησκευτικέ μειονότητες. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει αυτό. Αλλά κατόπιν πρέπει να βοηθήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας του IRA γιατί έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Ο κύριος Μπρόκ. Ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, Προεδρεύοντα, κύριε εκπρόσωπε, Νομίζω λοιπόν πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι η επίλυση του προβλήματος, το να, επέλθουν, ε, να επέλθει η σταθερότητα στη Λιβύη, αυτό είναι θέμα ανθρωπιάς για αυτή τη χώρα, αλλά είναι θέμα καθοριστικής σημασίας για μας. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε αυτή τη διαδικασία που ανέφερε ο συνάδελφος, θα πρέπει να τη συνεχίσουμε. Αυτό πρέπει να το πράξει η πατή εκπρόσωπος και τα κρατημέλη για να επιτύχουμε. Πρώτον, η αποστολή το μας ε, να δραστηριοποιηθεί, να ελέγχει τα χωρικά ύδατα και με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ε, διακινητές όσοι πράττουν λατρεμπόριο, γιατί αλλιώ μα περιμένουν πολύ χειρότερα ε, όσον αφορά την απόβαση των μεταναστών στην Ιταλία. Δεύτερον, πρέπει να επιτύχουμε τη σταθερότητα στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν είναι επιγόντω απαραίτητο να χορηγηθεί οικονομική βοήθεια, βοήθεια για τη σταθερότητα στη χώρα, να σταθεροποιηθεί η χώρα, έτσι ώστε να μπορεί και αυτή να εκπληρώσει τι εσωτερικέ τη υποχρεώσει. Γιατί και εδώ οφείλουμε να πούμε ότι τα κράτη-μέλη πολλά λένε και εύκολα λένε, αλλά κανεί δεν έχει καταβάλει τη εισφορά του στο καταπιτευσματικό ταμείο για την Αφρική. Να εκπληρώσουν λοιπόν τις υποχρεώσεις του τα κράτη-μέλη για να υπάρχει κάποιο περιθώριο να βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτή τη χώρα και να υπάρξουν εξελίξεις οι οποίες δεν θα επιτρέπουν να σταθεροποιηθεί, να πιάσει πόδι η ISIS, να βάλουν χέρι στις πετρελοπηγές και σε αυτές τις Αλγερίες, γιατί αν γίνουν όλα αυτά, να ξέρετε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα με μετά από αυτά που έγιναν στη Συρία και το Ιράκ. Και γι' αυτό όλα αυτά που σα λέω έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Ο κύριο Παντσέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η οι υποδείξεις στο σχέδιο ψηφίσματος είναι αρκετά σαφής. Ε, η πολιτική συμφωνία στη Λιβύη αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κατάσταση που δεν είναι πλέον βιώσιμη και να δημιουργήσουμε ένα ε, δημοκρατικό κράτος. Η συμφωνία στο Μαρόκο εγγυάται μια κυβέρνηση που θα βασίζεται στην αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών και θα ε, ενισχύσει τα θεσμικά όργανα, κυρίως την Εθνική Συμφωνία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει σε όλες τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Λιβύη. Καθήκον μας σήμερα είναι να εφαρμόσουμε όλες τις πολιτικές και διπλωματικές δράσεις ε, ώστε να εγκριθεί συμφωνία αλλά και να εφαρμοστεί και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες βάσεις για μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των ε, ενδιαφερομένων στη διαδικασία εθνική συμφιλίωσης. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να επισημάνω τρία στοιχεία πέραν των όσων ε, ήδη αναφέρονται στο ψήφισμα, τα οποία θα πρέπει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστούν περαιτέρω. Καταρχά, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο των γειτονικών χωρών. Ένα ρόλο ο οποίο ήδη διαδραματίζεται στη διαδικασία τη σταθεροποίηση και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το ρόλο. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας επεραιτέρω ρόλος που θα βοηθήσει ε, τους Δήμους ακριβώς για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει, ε, έχει δομηθεί η Λιβική κοινότητα των ε, φυλών και θα πρέπει να βοηθήσουμε τη διαδικασία αυτή τη δημοκρατική σταθεροποίηση. Τέλο, έναν περαιτέρω μήνυμα που πρέπει να αποστείλουμε εμεί από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να αποφύγουμε τα σφάλματα του παρελθόντο. Ε, η διεθνή κοινότητα και η άρχουσα τάξη θα πρέπει αυτή τη φορά να ε, χρησιμοποιήσει ε, μεγαλύτερη ταπεινοφροσύνη με ένα μακρόπνο όραμα και να χρησιμοποιήσει το μυαλό τη και όχι μόνο τα συμφέροντά του. Ο κ. Δεμεσμέκη, ένα λεπτό. Οι συζητήσεις για την ε, Λιβύη είναι συζητήσεις όπου βλέπουμε συνέχεια μια επανάληψη. Εξακολουθούν τα άτομα να λένε ότι τελειώνει ο χρόνος για τη, Λιβύη, για τη Υπάρχει ε, αναρχία, διαπερατά σύνορα, ένα τεράστιο και άπελπι πρόβλημα με τους πρόσφυγες και οι τρομοκράτες όλο έχουν και περισσότερο έδαφος που καταλαμβάνουν το Ισλαμικό κράτος ε, κερδίζει έδαφος όπως το Ιράκ και τη Συρία και αυτή τη στιγμή είναι 700 χιλιόμετρα η απόσταση που τους χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι μια μεγάλη απειλή για όλους μας. Στρατολογούν άτομα φτωχούς οι οποίοι δημιουργούν πολιτοφυλακές κάποιου είδους Χωρί καμία σταθερότητα στη Λιβύη, λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στη σύνολη περιοχή. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε να βρούμε μια περιεκτική και πλήρη συμφωνία. Μπορεί με μια συμφωνία ειρήνη να μπορέσει να ε, ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να σταθεροποιηθεί η εκεί, ίσω με τη βοήθεια τη Αφρικανική Ένωση. Αυτό λοιπόν είναι μια απαραίτητη προσπάθεια. Δεν έχετε άλλο χρόνο, κυρία Σπινέλη. Είμαι λιγότερο αισιόδοξο από σας κύριε Γκέπνερ. Μετά τον ιωστό πόλεμο στην Λιβύη γνωρίζουμε πια τις ε, επιπτώσεις του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Μην ξεχνάτε ότι οι πρόσφυγες είναι καρπός του χάους που σπίρουμε, σπέρνουμε εδώ και χρόνια παντού. Οι foreign fighters μιλούν ε, μπερδεμένα για το Ισλάν αλλά στο, τον εαυτό του τον βλέπουν σαν μια world generation. Δεν ξέρετε να λύσετε τον ε, γόδιο δεσμό της ε, Συρίας και σας επιβάλλουν τα δικτάτ οι Τούρκοι, δεν θέλουν τους Κούρδους. Η μόνη, ο μόνος που ίσως καταλαβαίνει την ε, αναγκαιότητα των Κούρδων είναι ο Πούτιν, αν θέλουμε να χτυπήσουμε την ίση. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λιβύη. Η αποτυχία του 2011 άνοιξε την πόρτα στο ISIS και τώρα η παρέμβαση που θέλουμε να κάνουμε γίνεται χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει κράτος στη Λιβύη. Επιπλέον η Ιταλία δεν πρέπει να πατήσει στη Λιβύη λόγω του, του απικιακού της παρελθόντος. Ευχαριστώ. Σεμπαστιά, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι προφανές ότι η Ένωση δεν έπαιξε πολύ καλό ρόλο στη Λιβύη. Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για το αν πρέπει να σταλούν στρατιωτικές δυνάμεις εκεί. Τι κάνουν οι χίλιοι ε, Βρετανοί 1500 Ιταλοί στρατιώτες πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον δύο στόχοι. Πρώτον, να έχουν εξαντληθεί με πάση θητεία η δινευτική διαδικασία η σύσταση μια κυβέρνηση εθνική ενότητα που εξυπηρετεί το, τα συμφέροντα του λαού τη Λιβύη. Δεύτερον, να βοηθήσουμε του πρόσφυγε που υποφέρουν ε, από τον πόλεμο, ε, απο, αποσταθεροποιώντα την ε, Μεσόγειο, ιδίω την, την Η λύση ωστόσο αυτή δεν μπορεί να είναι πλήρης αν δεν υπάρξει αναφορά και στον Περναντίνο Λεόν, τον είπα το εκπρόσωπο του ΟΗΕ που ταυτόχρονα διαπραγματεύεται στον, ε, στα πλαίσια του ΟΗΕ με μεγάλη εσωτερική εμπλοκή. Πρόκειται για μια σύγκρουση συμφερόντων που δεν μπορεί να μην, να συμπεριλαμβάνεται στο ψήφισμα αυτό. Κύριε Σεμπαστιά, δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Κάρβερ. A blue card Μπλε κάρτα είπαμε από τον κύριο Κάρβερ. Με χωρί μικρόφωνο κύριος Κάρβερ. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι που δέχεστε την μπλε κάρτα. Μπορείτε να συμφωνήσετε μαζί μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπλέκεται σε ακόμα περισσότερα περισσότερες δυσκολίες και περιπλέκει την κατάσταση. Μήπως θα πρέπει να αφήσουμε το θέμα αυτό στην Αφρικανική Ένωση με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναμειγνύεται κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση. Δεν συμμερίζομαι την άποψή σα, αγαπητέ συνάδελφοι. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να συμμετάσχει με στρατιωτικά μέσα. Αλλά είμαστε στα σύνορα της Συρίας. Έχουμε συμφέροντα για τα θέματα αυτά και έχουμε και μία έκκληση να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένω, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε το πρόβλημα της σύγκρουσης στην ε, Λιβύη. Ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα, ο Σφίντ. Ευχαριστώ η υποστήριξη του Κάμερον για, τον, για το ψήφισμα ε, είναι κλασικό παράδειγμα της κοντόφθαλμης αντίδρασης στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα ε, σήμερα και αντί για στρατηγική σκέψη έχουμε τέτοιες αντιδράσεις. Ε, με την ανατροπή μιας δικτατορίας δημιουργήσαμε αναρχία, αφήσαμε κενό εξουσίας που έδωσε τη δυνατότητα στο Ισλαμικό κράτος να εκμεταλλευτεί την κατάσταση που οδήγησε αυτό σε μια ανθρωπιστική κρίση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι συνέπειε, τι είδαμε και το καλοκαίρι και εξακολουθούμε να τι βλέπουμε στην Μεσόγειο, στη Σκανδιναβία, στο Καλέ και φυσικά στις πρόσφατες, στα πρόσφατα δρόμενα στη Γερμανία. Και τώρα θέλετε ε, στρατιωτική λύση. Ακούσαμε από τον πρόεδρο στην Επιτροπή Άμυνας ε, την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι τέτοιες αποστολές είναι καταδικασμένες ε, σε αποτυχία και αντί να κάνουμε τέτοιες αποστολές και να προωθούμε τέτοιες ε, στάσεις, ε, να σταματήσουμε και να μην κάνουμε δράσεις χωρίς σκεφτόμαστε τις συνέπειες. Έχετε μια μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Άκουσα πολύ προσεκτικά. Σας κατάλαβα καλά ότι κατά την άποψή σας ήταν λάθος στην στο να ε, συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανατροπή του Καντάφη στη Λιβύη. Ναι. Εάν παρεμβαίνει κανείς σε ξένες χώρες, χωρίς σχέδια, για να διορθώσει μια κατάσταση, αυτό που επιφέρει είναι φρίκη στο λαό της περιοχής και της χώρας, ε, δημιουργείς ε, το υπόβαθρο για την τρομοκρατία και μετά ε, οι συνέπειες βρίσκονται στα σύνορά σου. Ελπίζω να ήταν σαφές. Ένα λεπτό κύριε Ναούτου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κατάσταση στη Λιβύη, στη Λιβύη συγγνώμη, είναι αποτέλεσμα μεταξύ άλλων της παρέμβασης του Νικολά Σαρκοζή υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και που υποστήριξαν ορισμένοι ε, Γάλλοι σοσιαλιστές και γολικοί βουλευτές. Ε, ο μόνος που μπορούσε να εννοποιήσει τις περίπου 150 φυλές που ζούσαν στη Λιβύη ήταν ο, Κα, ο Καντάφη και κατάφερε να το κάνει με πολύ χαμηλό ε, πληθωρισμό και ανεργία. Αυτό καταστράφηκε τώρα. Η λύση θα ήταν να καλέσουμε τις φυλές που είναι αντίθετες με, την, με το Ισλαμικό κράτος. Είχα συζητήσει στη Ρώμη με τον Φράνκο Ρομπέρτη υπεύθυνο κατά της ε, μάχης τη Μασία που μου είπε τα εξή ότι φοβούνται ότι οι ομάδες, οι ομάδες Ισλαμιστών εμπλέκονται στην διακίνηση μεταναστών. Δεύτερον, μεταξύ των μεταναστών ε, μας είπε θα υπήρχαν σίγουρα τρομοκράτες που συνδέονται με το Ισλαμικό κράτος. Ξέρουμε ότι ο ε, προχωρά στη Λιβύη και αυτό δημιουργεί φόβους για την δική μας ασφάλεια πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτές τις ενοποιητικές στάσεις που κυριαρχούν εδώ και να σταματήσουμε την παράνομη μετακίνηση από τη Λιβύη. Σοπράδια, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση στη Λιβύη είναι κάτι περισσότερο από ανησυχητική. Μα υπόσχεται ένα πολύ ζωφερό μέλλον στην Ευρώπη αν δεν δράσουμε ταχαίω. Οι επιθέσει του Ισλαμικού κράτου κατά των τερματικών σταθμών στην Ανατολική Σύρτη, η κατάσταση τη πόλης της Ούν στο Θεζά. Όλες αυτές οι επιθέσεις του Ντάς, του Ισλαμικού κράτους, δείχνουν ότι ο εχθρός κερδίζει έδαφος. Υπάρχουν δύο θεμητοί λόγοι για να παίρνουμε στη Λιβύη. Καταρχήν για να αναχαιτήσουμε την ταχεία προέλαση του Ισλαμικού κράτους και δεύτερον την έκρηξη στις ροές παράνομων μεταναστών η παρέμβαση εναντίον του Καταφή έχει ανοίξει τους εσχώς του αιώλου. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι ταχαίως για να έχουμε δύο βασικές λύσεις. Πρώτα μια ευρωπαϊκή στρατιωτική ε, επιχείρηση μαζί με την Αίγυπτο για να εξαλείψουμε το Ισλαμικό κράτος. Η Γαλλία όμως δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Και δεύτερον, να δημιουργηθούν κέντρα κράτησης και διαλογής για τους ε, υποψήφιους πολιτικής πρόσφυγες από την ε, Λιβύη και από όλους αυτούς που έρχονται και περνούν από τη Λιβύη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το κάνουμε και χρειαζόμαστε και τη βοήθεια ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας. Ένα λεπτό και τριάντα κύριε Σπρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν παρατηρεί κανείς τη Λιβύη, έχει μια εντύπωση déjà vu, ότι είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί. Για μια ακόμα φορά βρισκόμαστε σε απόλυτο αδιέξοδο η συμφωνία του Τομπρούκ, η κυβέρνηση του Τομπρούκ παρά το γεγονό ότι είχε αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα, έχει απορρίψει την κυβέρνηση του, που δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Παρά την συμφωνία την πολιτική που επετέφθη τον προηγούμενο Δεκέμβριο, έχει διαλυθεί και η τελευταία ελπίδα για σταθερότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει αυτή η συμφωνία να πάρει σάρκα και ουστά, να μπορέσει να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη κυβέρνηση Εθνική Ενότητα, η οποία να θεωρείται νόμιμη από του Λίβιου. Όσο δεν γίνεται κάτι τέτοιο, όσο δεν μπορεί να υπάρξει κάποια συμφωνία, το Ισλαμικό κράτο εκμεταλλεύεται αυτήν την αστάθεια και κερδίζει περισσότερο έδαφο. Αυτό ο τρομοκρατικό φορέα απειλεί όχι μόνο την ασφάλεια τη Λιβύη, αλλά επίση και την οικονομική επιβίωση τη Λιβύη επιτίθεται κατά των πετρελαϊκών υποδομών και θέτει σε κίνδυνο τη μόνη πηγή εσόδων της Λιβύης η οποία βρίσκεται σε μια καταστροφική οικονομική κατάσταση. Θα πρέπει προφανώς να ακολουθήσουμε τους διπλωματικούς δρόμους για να επιλύσουμε την <clears throat> ε, κατάσταση στη Λιβύη αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ανάγκη στρατιωτικής παρέμβασης. Η κυβέρνηση της Λιβύης όμως δεν μπορεί να ζητήσει τη βοήθειά μας εάν δεν υπάρχει. Μια στρατιωτική λοιπόν ε, παρέμβαση από την Συμμαχία μπορεί να γίνει μόνο μαζί με μια αποτελεσματική πολιτική στρατηγική που να είναι αποδεκτή από όλου του λίδου. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε για να μπορέσουμε να καθορίσουμε αυτή τη στρατηγική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η δύο λεπτά. Η Ευρωπαϊκή... Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη απέτυχαν να έχουν μια συνεκτική στα στρατηγική για να μπορέσει να υπάρξει μια μετάβαση στη Λιβύη. Χωρί μια τέτοια στρατηγική είναι πολύ φανερό ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία κυβέρνηση, δεν θα μπορούν να υπάρχουν δυνάμεις ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο, δεν μπορεί να υπάρξει παροπλισμός των πολιτοφυλακών, δεν μπορεί να υπάρξει αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων και των τρομοκρατών που χρησιμοποιούν τα εγκαταλελειμμένα οπλοστάσια που έρχονται από χώρε όπω είναι η Γυρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατη εξακολουθούν κάθε φορά να αφήνουν τις, τους φιλετικές αντιπαραθέσεις να έχουν το πάνω χέρι στην ε, Λιβύη και γίνεται ένας αγώνας ε, αντιπροσώπων μεταξύ Σουνιτών και Σιητών που χρηματοδοτεί και με τη Σαουδική Αραβία που υποστηρίζει τους αλαφίστες ενώ η Τουρκία και άλλες χώρες υποστηρίζουν τους αδερφούς μουσουλμάνους. Με τον τρόπο αυτό έχει διαλυθεί η Λιβύη και είναι έφορο έδαφος για τους ε, τρομοκράτες η προσπάθεια για μια συμφωνία στη Λιβύη μα δίνει μια ευκαιρία η οποία μπορεί να βοηθήσει τη Λιβύη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη την περιοχή να μην βρεθούν σε απόλυτο αδιέξοδο. Είναι η τελευταία ευκαιρία για να μπορέσουμε να εμποδίσουμε την κλιμάκωση τη βία. Η τρομοκρατική επίθεση που οργανώνεται από τη Λιβύη στην Ευρώπη είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα. Κανεί λοιπόν δεν θα πρέπει να αποκλείσει τη δυνατότητα μια πολιτικής, παρέμβαση. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η κυβέρνηση θα μπορέσει να επιβάλλει τη θέλησή τη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει <clears throat> να επιβάλλει κυρώσει εναντίον οποιασδήποτε οργάνωση ή ατόμου που δεν υποστηρίζει αυτή τη συμφωνία. Η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να προασπίσει τα ζωτικά συμφέροντα της με την ασφάλεια στην Λιβύη. Ο αγώνας κατά των τρομοκρατών σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν οι πολιτοφυλακές, να σταματήσει το λαθρεμπόριο ανθρώπων και όπλων και να υπάρξει ενιαία διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων της ε, Λιβύης. Αλλιώς δεν θα υπάρξει ποτέ ασφάλεια, κυβέρνηση μετάβαση, σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έλεγχος των πετρελαϊκών πόρων και των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει για τη δική της ασφάλεια και την ασφάλεια της περιοχής. Η κυρία Φωτίγκα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη θα δημιουργηθεί γρήγορα γιατί είναι αναγκαίο για την ασφάλεια του πληθυσμού, την καταπολέμηση του ΝΤΑΕΣ και την άντληση των ξένων ε, των διεθνών πόρων. Χρειάζεται ταυτόχρονα να υπάρξει έλεγχος της παραγωγής πετρελαίου. Υποστηρίζω την ε, τις προσπάθειες της ΥΠΑ εκπροσώπου και της διεθνούς κοινότητας. ο κύριος Αλιώ, ένα λεπτό. Συνάδελφοι, εδώ μας οδηγούν οι περιπέτειες που είχε υποστήριξει μια σειρά βουλευτών εδώ, περιπέτειες του κύριου Σερκοζή Παγιού, ε, προέδρου της ε, ε, Γαλλίας και του ψευτοφιλόσοφου κυρίου Μπερνάρ Ανρί Λεβί. Η κατάσταση στην Λιβύη είναι άμεσο αποτέλεσμα της περιπέτειας στην Λιβύη. Η κυβέρνηση, αυτή είναι η πραγματικότητα, σήμερα μιλά με τρομοκράτες. Οι Ισλαμιστές ή όχι, αλλά τρομοκράτες. Κανείς δεν θέλει να συζητήσει. Συνεχίζουμε να συζητάμε με το κοινοβούλιο του τον Μπρουκ που είναι το κλειδί εν μέρη της αποκατάστασης σε αυτό το γεωπολιτικό εγκληματικό χάος που δημιουργήσαμε, μια αποστολή ευρωβουλευτών στο Μαλί πήγε για να δει την κατάσταση. Δεν μπορεί να κάνει λάθος πια για το ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι αντίπαλοι μας στην περιοχή. Ο κύριος Μίλαν μόνο 1,5 λεπτό η πολιτική συμφωνία ε, του περασμένου Δεκεμβρίου στην Σχήρα και που υποστήριξε εν μέρει από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 22 στο 2259 ψήφισμα ήταν θετικό για την Λιβύη ε, που εγκρίθηκε και από το κοινοβούλιο του Τόμπρουκ ε, την περασμένη εβδομάδα. Αυτό απορρίπτει το ΑΘΟΚ αυτό και η απόρριψη του άρθρου 8 είναι μεγάλα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν το συντομότερο δυνατό η πολιτική διάσταση επιδίνωσε την η πολιτική... το πολιτικό χάος επιδίνωσε την οικονομική... Ε, το οικονομικό χάος που δημιουργεί σοβαρή ανησυχία. Το Ντάες φαίνεται ισχυρό στη Σύρτη και είδαμε την ικανότητα που έχει να αποσταθεροποιεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Χρειαζόμαστε μια οριστική συμφωνία η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το συντομότερο δυνατό. Αυτό θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να χτυπήσουμε τον ΤΑΕΣ και να ηρεμήσει και να ειρηνεύσει η Λιβύη, η χώρα που έχει επιπτώσεις στους γειτονές της, την Αίγυπτο, την Τινησία και την Αλγερία. Ταυτόχρονα η Λιβύη συνδέει άμεσα την Μεσόγειο με το Σαχέλ. Ε, είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει ταχύτατα κυβέρνηση εθνικής ενότητας που θα χτυπήσει την δημοκρατία και τη διακίνηση ανθρώπων για να οδηγήσει την Λιβύη στην ειρήνη και την ευημερία. Ελπίζω και ο Σκόπλερ, υπεύθυνο ε, και ο ΙΕ να μπορέσουν να συμβάλλουν σε μια γρήγορη υπέρβαση των υφισταμένων εμποδίων. Ο κύριος Παρινιέ, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά τις συζητήσεις, ε, μετά τον προβληματισμό πρέπει να περάσουμε στη δράση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το χάος ε, που διαπιστώνουμε στη Λιβύη αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις απειλές στην Τινησία και τις απειλές που δέχεται η Ευρώπη θα πρέπει να δράσουμε. Και αυτό ζητώ από τις Ευρωπαϊκές Αρχές, από το Συμβούλιο και από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο. Καταρχάς, θα πρέπει στρατιωτική στρατιωτικές κινήσεις ε, να δρομολογηθούν. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ε, μια κυβέρνηση εθνική ενότητα και κράτο δικαίου. Και θα πρέπει να πούμε στην, ε, στο κοινοβούλιο του τον να δεχτούν την κυβέρνηση εθνική ενότητα, ούτω ώστε να επιτρέψουμε τι ε, στρατιωτικές επιθέσεις και την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους. Θα πρέπει βεβαίως να καταπολεμήσουμε τη μαφία, τους διακινητές ανθρώπων που προκαλούν και σπέρνουν θάνατο. Φυσικά θα πρέπει να δώσουμε οικονομική βοήθεια με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσουμε τους κατοίκους κλειδίς. Ευχαριστώ. Υπάρχει μία μπλε κάρτα. Το τι δέχεστε. Τι δέχεστε. Να ζητήσω, να ρωτήσω το συνάδελφο αν συμφωνεί όπως ζητάει η κυβέρνηση των Μπρουκ να αρθεί το εμπάργο. Χωρίς το εμπάργο λέει ότι μπορούμε να βρούμε πιο γρήγορες λύσεις. Ανταυτού η κυβέρνηση του τον Μπρουκ λόγω του εμπάργου δεν μπορεί να κάνει αυτά που θα ήθελε να κάνει. Ενώ οι αδερφοί μουσουλμάνοι έχουν την δυνατότητα υποτίθεται να κάνουν αυτά που θέλουν. Για να απαντήσω στο ερώτημα Σήμερα πρέπει οι γείτονες, η Αίγυπτος, αλλά και η Αλγερία, το Μαρόκο και την Ισία να συμμετάσχουν σε μία συζήτηση μαζί με το Κοινοβούλιο του Τομπρούκ, ούτω ώστε να βρεθούν διπλωματικέ λύσεις. Και αυτή η συμφωνία του Κοινοβουλίου του Τομπρούκ να επιτρέψει να δημιουργηθεί αυτή η κυβέρνηση εθνική ενότητα, Το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ή όχι το εμπάργο. Το βασικό είναι να βρούμε μία λύση, ούτω ώστε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το Ισλαμικό κράτος. Ο κύριος Μπέλντερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. οχι το εμπαργκο το βασικο ειναι Προεδρία, κύριε Κούντερες, έχει ήδη Έχω εκτιμήσει πάρα πολύ την παρουσία σας εδώ και κύριε Πρόεδρε είναι πάρα πολύ σαφές ότι η Λιβύη γίνεται πεδίο μάχης για το Ισλαμικό κράτος. Και έχουν πια το ορμητήριό τους εκεί. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί στόχος του Ισλαμικού κράτους εκεί. Είναι πολλά από τα λιμάνια της Λιβύης που αυτή τη στιγμή έχουν καταληφθεί από το Ισλαμικό κράτος. Η Λιβύη είναι μια άμεση απειλή για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όπως είπε ο κύριος Υπουργός Κιόντερς, εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Αλκάιντε, του αδελφούς μουσουλμάνους και το Ισλαμικό κράτος και θα να ξέρω την άποψή για το θέμα αυτό. Ο κύριο Κούκαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Διακεκριμένοι συνάδελφοι, εγώ θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια στη Λιβύη να επιτυχούν μια πολιτική συμφωνία για να υπάρξει η δημιουργία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική τομή και πρόοδο για την Λιβύη για να επιτευχθεί η σταθερότητα και η ειρήνευση στην περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι μια τέτοια λύση θα γίνει πραγματικότητα. Μόνο μια ενωμένη Λιβύη μπορεί να αντιμετωπίσει την διαδικασία, τη δύσκολη διαδικασία του να οικοδομήσει ασφάλεια και οικονομική ευμάρεια. <clears throat> Το συνεχιζόμενο χάος στην Λιβύη είναι μια απειλή για την ε, ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί μπορεί να δώσει λαβή σε, μια νέα, σε ένα νέο κύμα προσφύγων. Γι' αυτό υποστήριξε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειρήνη στη Λιβύη και όλους τους νότιους γείτονές μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να είναι ένας σημαντικός ε, βοηθός για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης να ενισχύσει το τομέα ασφαλείας της Λιβύης. Ας τονίσουμε στους Λίβιους ότι είμαστε μαζί τους. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριε Βαλενθιάνο. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τους διαπραγματευτές για αυτό το ξεκίνημα συμφωνίες. Θα ασχοληθώ στο λίγο χρόνο που έχω ζητώντας βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λιβύη. Δεν παρέχεται η βοήθεια που απαιτεί το πρόγραμμα ανθρωπιστικής ανταπόκρισης. Χρειάζεται βοήθεια 1,5 εκατομμύρια άτομα. Η ανθρωπιστική δράση δεν είναι πολιτική, αλλά για να το πετύχει, για να πετύχει πολιτική λύση πρέπει να λύσει την ανθρωπιστική κρίση. Αυτό το χειμώνα πολλοί άνθρωποι χρειάζονται επιγόντω την παρέμβασή μας. Απευθύνω έκκληση λοιπόν στους υπεύθυνους της Επιτροπής, τις υπηρεσίες μας, τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής της Εξωτερική Δράσης να έχουν επίγνωση ότι μόνο, η πολιτική, μόνο μια πολιτική συμφωνία δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να ζήσει. Θέλει ρούχα ο άνθρωπο, θέλει βοήθεια, θέλει φαγητό, θέλει διέξοδο που θα του δίνει έναν ορίζοντα Σε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπασίρ, ένα λεπτό. Υποστηρίζω τις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και ελπίζω ότι θα φέρουν διαρκή ειρήνη στη Λιβύη. Η πραγματικότητα επιτόπου είναι πολύ ανισχυτική. Όλο και περισσότερες κατολογίε για επερχόμενη στρατιωτική επέμβαση στην Λιβύη δείχνουν ότι η χώρα είναι πολύ κοντύτερα στο χάος παρά σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ένα κατηγορό για την ανικανότητα της διεθνούς κοινότητας να επιφέρει θετική αλλαγή στην περιοχή. Αν η Λίμπια ε, διαλυόταν ξανά, αυτό θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην Τινησία. Δυστυχώς είναι το μόνο, η μόνη ελπίδα ε, που απέμεινε από τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Αυτό θα επιτείνει την, κατα τη ζωφερή κατάσταση και θα έχει άσχημες συνέπειες. Θα πρέπει να βρούμε ε, λύσεις με τους Λίβιους για τα λιβικά προβλήματα. Αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί αν αποτύχουμε ακόμα μια φορά, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δραματικά από, από αυτά που ζουν τώρα οι Λίβοι. Ο κ. Μακάλιστερ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με αυτό το ψήφισμα για την κατάσταση στη Λιβύη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιστεί την, εφιστά την προσοχή σε μια χώρα που βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Όπως ακούσαμε σήμερα, η ανθρωπιστική κρίση στη χώρα επιδεινώνεται. Εξτεμιστικές οργανώσεις και κινήματα στη Λιβύη είναι όλο και περισσότερα και δημιουργούν μείζονες απειλές στην σταθερότητα όλης της περιοχή ε, σε γειτονικέ χώρες όπως ε, η Αίγυπτος και κυρίως η Τινησία ε, κινδυνεύουν ότι η κατάσταση ανασφάλειας θα φτάσει και εκεί. Θα πρέπει η Λιβύη να επωφεληθεί από μια κατάσταση ασφάλειας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε. Ε, μια αρχική ε, κατάπαυση του πυρός και ένας μηχανισμός παρακολούθησης θα ήταν σημαντικό. Αυτές οι δράσεις όμως ε, δεν έχουν και πολλέ πιθανότητες επιτυχίας εάν δεν επικυρωθούν από την κυβέρνηση και αν δεν υπάρξει κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίζει τη Λιβύη για να κάνει αυτό το μείζον βήμα δημιουργία αυτή τη κυβέρνηση. Η κατάσταση στη Λιβύη γίνεται απελπιστική οι εξτρεμιστές του ΝΤΑΕΣ επεκτείνονται. Πρέπει να τους σταματήσουμε τώρα. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να περιμένει την διαμόρφωση κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για να μπορεί να υπάρξει σεβασμός από πλευράς του, του λαού της Λιβύης. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσει είχαν προβλήματα, γιατί υπάρχουν σαφείς ε, το, μέσα στην λιβική κοινωνία. Δεν μας εκπλήσει η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, ούτε θα έπρεπε να γνωρίσουμε τα λάθη στις ε, προσπάθειες διαμεσολάβησης. Οι βασικοί δρόντες ε, στην Λιβύη έχουν αντιφατικά συμφέροντα και προοπτικές. Είτε είναι καλόπιστοι είτε είναι κακόπιστοι πρέπει να αποφασίζουν για το μέλλον του λαού τους. Η επιβολή κυρώσεων στη ενόψη της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας είναι λάθος μήνυμα, ιδίως αν γίνει εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ. Δημιουργώντας, δημιουργεί κάτι τέτοιο ε, κακή αντιμετώπιση της Ευρώπης και ενισχύει τον ΤΑΕΣ. Πρέπει να διαμορφώσουμε μια εθνική διοίκηση, το οποίο είναι επικίνδυνο, αλλά είναι μία από τις επικίνδυνες λύσεις. Ο κύριος Πιωτρόφσκι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και τέσσερα χρόνια παρακολουθούμε από την Ευρώπη τα γεγονότα στη Λιβύη. Και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην κατάσταση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τροφοδοσίας με πετρέλαιο και άλλες απειλές. Έχουμε δύο <clears throat> κοινοβούλια στη Λιβύη που σχεδόν κατάφεραν να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με βάση τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν μια θετική συνεργασία, υποστηρίζεται επίσης και από τη δική μας ε, ομάδα. Θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτή τη λύση και να θυμηθούμε ότι με την ε, συμφιλίωση των δύο αυτών αντίμαχων πλευρών δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια τρίτη δύναμη και δεν πρέπει να ενισχύσουμε τους εξτρεμιστές του Ισλαμικού <clears throat> κράτους που εξακολουθούν να καταδιώκουν τους χριστιανούς στη χώρα αυτή. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους σταματήσουμε. Ο κύριος Φίσας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όπως έχω πει πολλές φορές σε αυτή την Ολομέλεια, η πάρα πολύ μεγάλη εξουσία του Καντάφη στη Λιβύη στο παρελθόν οδήγησε σε ένα αποτυχημένο κράτος στην Λιβύη γιατί οι εξοπλισμοί που είχε στα χέρια του οδήγησαν στην πιο εύκολη αποσταθεροποίηση της Λιβύης και όπως είπε ο πρόεδρος Μπουχάρη σήμερα η Νότια Λιβύη είναι ε, μια τεράστια αγορά όπλων. Η Λιβύη αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, την ε, προέλαση <clears throat> του Ισλαμικού κράτους, τα προβλήματα στις πετρελαϊκές υποδομές και επίσης μια καταστροφική οικονομική κατάσταση λόγω της μεγάλης της εξάρτησης από το πετρέλαιο το οποίο έχει καταρρεύσει τη τιμή. Ενώ αυτής της κατάστασης λοιπόν μιας χώρας που βρίσκεται στις θύρες της Ευρώπης είναι απαραίτητο να κάνουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε να εφαρμοστεί η πολιτική συμφωνία που ε, υπεγράφει τον προηγούμενο Δεκέμβρη και κυρίως να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος με έδρα στην Τριπολίτη. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριο Καν. Πρόεδρε, δεν έχουμε πια χρόνο για να σταθεροποιήσουμε τη Λιβύη. Η ανθρωπιστική βοήθεια, η, ασφάλ... η κατάσταση ασφάλειας είναι τρομακτική. Ο ΆΙΣΙΣ ανεβαίνεται και έχει πρόσβαση σε πετρελαϊκές ε, πηγές. Οι Αμερικανοί προσπαθούν με στρατιωτικές επιλογές να σταματήσουν την προέλαση του ISIS η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίξαμε με ανθρωπιστική βοήθεια τη Λιβύη και με βοήθεια στην πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Οι Λίβοι θέλουν να επιτύχει αυτή η συμφωνία μετά από πέντε δύσκολα χρόνια. Θέλουν κάποια ελπίδα. Μόνο μια κυβέρνηση εθνική συμφωνία μπορεί να σταθεροποιήσει τη Λιβύη. Το Κοινοβούλιο τη Λιβύη πρέπει να εξασφαλίσει ότι ότι παρότι είναι τέλεια αυτή η συμφωνία για την κυβέρνηση Εθνικής Συνότητα, πρέπει να επικυρωθεί ούτω ώστε η κατάσταση στη Λιβύη να μην γίνει απελπιστική. Εμεί θα πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη ανθρωπιστική και αντεξιακή βοήθεια. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε άλλον στρατιωτικό ηγέτη να χρησιμοποιήσει την ε, Λιβύη, ε, γιατί δεν χρειάζεται άλλο καντάφι η Λιβύη. Ζητάσκα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Λιβύη βρίσκεται 200 μόνο χιλιόμετρα από την Ευρώπη. Πέντε χρόνια μετά την πτώση του καθεστώτος Καβάφη, ε, βρίσκεται σε χάος. Είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση Εθνική Ενότητα και να αναχαιτήσουμε την προέλαση του Ισλαμικού κράτους, το οποίο έχει καταλάβει δηληστήρια και αυτή τη στιγμή ενισχύει τη θέση του υπέρ της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να υπάρχει η παράνομη λαθρεμπορία όπλων και η λαθρεμπορία ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Όλο και περισσότερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων ζουν σε άθλιες συνθήκες. Γι' αυτό πρέπει η Λιβύη να έχει μια σαφή αντιμετώπιση από τις πολιτικές ελίτ και η Ευρώπη πρέπει να δώσει την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια. Η κατεύθυνση στην οποία πηγαίνει η χώρα αυτή μπορεί να επηρεάσει όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Είπα καβάφι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Λιβύη είναι η γειτονική χώρα μας. Η κατάσταση είναι πολύ δραματική. Λόγω του πολιτικού κενού που υπάρχει, την εκμεταλλεύεται το Ισλαμικό κράτος και άλλες εξτρεμιστικές δυνάμεις. Η κατάσταση ανασφάλειας ε, επεκτείνεται στην Αίγυπτο, στην Τινησία, στις χώρες της Αχέλ, ακόμα και στην Ευρώπη. Στην άλλη όχθη της Μεσογείου εκτιμάται ότι υπάρχουν 3.000 μαχητές του Ισλαμικού κράτους. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρώσει πολιτικές προσπάθειες ε, στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Δεκεμβρίου ε, του 2015 για κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Αλλά αν δεν αποτύχει, θα πρέπει να εξετάσουμε και μια εναλλακτική λύση. Στρατιωτική επέμβαση από μια διεθνή δύναμη με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εμποδίσουμε να, την κατάληψη εξουσίας ε, στη Λιβύη από το Ισλαμικό κράτος. Η Λιβύη μην ξεχνάμε ότι είναι γειτονική χώρα πάνω απ' όλα. Μικρόφωνο παρακαλώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, την πεσμένη εβδομάδα δεν έγινε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό κακό νέο. Η απουσία κυβέρνησης αποσταθεροποιεί, όλη την περιοχή ενώ επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση αποσταθεροποιώντας και τις γειτονικές χώρες, την Ισία και την Αίγυπτο κυρίως. Το κενό στη Λιβύη είναι πρόσφορο έδαφος για τρομοκρατικές οργανώσεις όπως την ίσης. Η... Όσο δεν υπάρχει νόμιμη κυβέρνηση, οι ευρωπαϊκές δράσεις κατά της, ε, των διακινητών δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Μόνο μια νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης μπορεί να επιτρέπει στα σκάφη να μπαίνουν στα χωρικά της ίδρυτα. Γι' αυτό ζητώ από την Ένωση και τη διεθνή κοινότητα να κάνουν ό,τι μπορούν για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην χώρα. Η διαδικασία κατσιδιάει τώρα. Πέντε συνάδελφοι θα μιλήσουν, έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Πόσπισελ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουγα τη συζήτηση προσεκτικά. Συμφωνώ με την ανάλυση των συναδέλφων η κατάσταση είναι απελπιστική. Η Ευρώπη έχει μια σειρά μεταναστευτικών ροών, άλλων μεταναστευτικών ροών. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι που ήδη αναφέρθηκε. Οι απειλές για απαγωγή Ευρωπαίων πολιτών στην, στο έδαφος της Λιβύης. Να πω στους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής ότι πριν τον Μάρτιο του 2015 απήχθη ένας Τσέχος πολίτης, ο Μπάμπαλ Χρούζα, ο οποίος δούλευε σε μια πετρελαϊκή εταιρεία και είναι ένα χρόνο σχεδόν στα χέρια των τρομοκρατών. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν διαπραγματευόμαστε με τις τρομοκρατικές ομάδες. Ο κ. Μαριάς η τρέχουσα οικονομική και πολιτική αποσύνθεση της λιβύης πλήττει τον ήδη καταπιεσμένο λαό της χώρας. αρχικά παρατηρούμε ακόμη και σήμερα επιθέσεις εναντίον σημαντικών πετρελαϊκών υποδομών οι οποίες έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την ευημερία του πληθυσμού της λιβύης αφού το 80% του αεπ της εξαρτάται από τον πετρελαϊκό τομέα. πρόσφατα οι τρομοκράτες του νταές οι οποίοι έχουν εδραιώσει την επιρροή τους στη χώρα μετά την ανατροπή του καντάφη το 2011, συνέχισαν για δεύτερη μέρα τον βομβαρδισμό του λιμανικού αλλά και πετρελαϊκού σταθμού σταθμού sider προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου. αποτέλεσμα αυτής της εμπόλεμης κατάστασης στη λιβύη είναι ο εξαναγκασμός χιλιάδων ανθρώπων να εγκαταλείψουν τη χώρα εντείνοντας έτσι τις μεταναστευτικές ροές επομένως είναι σαφές ότι όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης θα πρέπει να αντιταχθούν στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που παρατηρούνται καθημερινά στη χώρα καθώς και σε κάθε ενέργεια που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. ταυτόχρονα πρέπει να στυλιτευτεί η δράση της τουρκίας που στηρίζει τους ντομποκράτες του Νταε που δραστηριοποιούνται στη λιβύη. ευχαριστώ. Όταν μίλησα σε αυτό το κοινοβούλιο για πρώτη φορά για τη Λιβύη, είπα ότι ξέρουμε τι δεν θέλουμε. Δεν θέλαμε τον δικτάτορα Καντάφη, θέλουμε μια δημοκρατική Λιβύη. Όμως δεν ξέρουμε πώς θα την πετύχουμε. Τώρα ξέρουμε τι θέλουμε και πώς θα το πετύχουμε. Γιατί είναι ασύλληπτο που κάμια δυο χιλιάδες ε, μαχητές δημιουργούν τέτοια προβλήματα στην άμεση γειτονία μας που αποσταθεροποιούν φιλικές χώρες και εμείς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Θα μπορούσαμε στο παρελθόν εμείς να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είναι κρίμα που δεν έχουμε τη διπλωματική δύναμη να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, γιατί χρειαζόμαστε επιγόντως να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Και ο Πόρτο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Λιβύη είναι ένα κενό ασφάλειας, ένα κενό εξουσίας, το οποίο ουσιαστικά καλύπτεται τώρα από το Ισλαμικό κράτος. Εμείς θα αποτύχουμε και πάλι να αφήσουμε τη Λιβύη στη δική της τύχη. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση όπλων φαίνεται ότι είναι πια το έδαφος της Λιβύης αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας Ακούσαμε και πολλές προτάσεις σε αυτή τη σημερινή συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εκπρόσωπος συγκεκριμένα του Συμβουλίου θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο. Γιατί πολλοί θέλουν να αφήσουν τη Λιβύη όπως είναι και αυτό δεν είναι προς το συμφέρον μας. Ευχαριστώ. Το να υποστηρίξουμε <clears throat> την ε, ανατροπή του Καντάφη από την Ευρώπη και την Αμερική μπορεί να ήταν σωστό, αλλά έπρεπε να δώσουν βοήθεια στη Λιβύη μετά από την ανατροπή του Καντάφη. Βλέπουμε ότι η χώρα αυτή μετά από 42 χρόνια δικτατορίας είναι πλέον σε ένα χάος. Τέσσερα χρόνια αργότερα μετά από την πτώση του Καντάφη δεν έχει σταματήσει ο εμφύλιος πόλεμος. Κανένα δεν πρέπει να εκπλήξει κάτι τέτοιο. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν κερδίσει έδαφος και πετρελαϊκές υποδομές σε μια χώρα με διαπερατά σύνορα, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το Ισλαμικό κράτο. Θα δρέψουμε του καρπού τη Αδράνεια μα μέχρι στιγμή, εάν δεν κάνουμε την απαραίτητη προσπάθεια να δώσουμε πολιτική, στρατιωτική και οικονομική βοήθεια για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τη δημιουργία μια λειτουργική και περιεκτική κυβέρνηση, η οποία θα ενισχύσει τη χώρα και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το Ισλαμικό κράτο. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο. Έχει κλείσει η διαδικασία Catch the Eye. Και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον Υπουργό, τον κύριο Κούντερς. Uh, uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση, για τις σημαντικές σας παρατηρήσεις. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, και εδώ μιλώ εκ μέρους είπα της εκπροσώπου, ότι η Λιβύη είναι κρίσιμο κράτος για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Είναι γειτονική χώρα. Ε, είναι κοντά στην Τινησία και στην Αίγυπτο, κοντά στο Μαλί και στο Νίγηρα και συμφωνώ με σας που είπατε ότι υπάρχουν κίνδυνοι, όλο ένα και αυξανόμενοι, παρουσίας του ισταμικού κράτους ε, στη Λιβύη. Η πολιτική διαδικασία, παρότι προχωράει επίσης, δεν προχωράει αρκετά γρήγορα. Υπάρχουν άπειρα εμπόδια και οι νέες αρχές είναι πολύ ευάλωτες, χρειάζονται την υποστήριξή μας. Συμφωνούμε, αν ακούσουμε προσεκτικά τα όσα είπαν οι προβουλευτές, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι τόσο κοντά στη Λιβύη αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές. Τρομοκρατικές ομάδες ενισχύονται, θα πρέπει να ανασχεθούν ο ISIS έχει δημιουργεί τεράστιες ε, απειλές στην, ε, στους πετρελαϊκούς πόρους της Λιβύης και είναι και όλο και πιο επίγον το να βρούμε πολιτικές λύσεις μέσω της ε, εφαρμογής της συμφωνίας και να επιτρέψουμε στις λιβικές δυνάμεις να ενωθούν κατά του ISIS και η λιβική οικονομία και ο κοινωνικός ιστός επειδή βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και υπάρχει σοβαρότατη ανθρωπιστική κρίση όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι διακινητές θα πρέπει να τιμεστούν και η λαθομετανάστευση θα πρέπει να ελεγχθεί. Σημαντικό επίσης να πούμε ότι όλοι ξέρουμε ότι η πραγματική λύση σε αυτά τα τρομακτικά προβλήματα θα ήταν μια λιβική κυβέρνηση που δέχονται όλοι οι Λίβοι και που θα τους εκπροσωπεί όλους και που θα υποφελείται από την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Ακούσα μια ερώτηση. Αν κοιτάξουμε τις διάφορες, τους διάφορους φορείς τις ε, πολιτοφυλακές, την παρουσία του Άισι σε τόσα πολλά σημεία της χώρας, είναι δυνατόν να υπάρξει συμβασμός. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν αμφιβάλλουμε ότι περισσότεροι Λίβοι δεν είναι εξτρεμιστές και δεν υπέρ του Άισις. Σε καμία, υπό καμία μορφή ή μόρφωμα. Οι νέες αρχές είναι σχετικά μετριοπαθείς και εκπροσωπούν τους μετριοπαθείς ε, Λίβιους. Και έχουμε την υποχρέωση να τους υποστηρίξουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί για να συνεισφέρει στις προσπάθειες αυτές, ούτως ώστε η Λιβύη να γίνει μετά από πέντε χρόνια απογοητεύσεων μια ασφαλής χώρα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι καταλαβαίνω γιατί πολλοί από σας θέλετε και ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αλλά πιστεύω και το πιστεύει και η διεθνή κοινότητα, ότι μία ε, κυβέρνηση εθνική Ενότητα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, που θα την ε, αποδέχονται όλοι οι Λίβοι ε, μετά από διαπραγματεύσει, είναι η μόνη περίπτωση για να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η ειρήνη και στην περιοχή και να αποφευθεί οικονομική κατάρρευση. Δεν είναι αφέλει αυτό. Το πιστεύει. Ε, και αυτό και η εκπρόσωπος δεν πιστεύω ότι η στρατιωτική λύση είναι η πιο σοφόνος λύση. Φυσικά θέλουμε να υποστηρίξουμε τις διαπραγματεύσει. Είπατε εκπρο... εκπρόσωπο είναι ενεργή. Ε, συνεργάζομαστε με τον Μάρτιν Κιούμπλερ και θέλουμε να χειροκροτήσουμε τη δουλειά του μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τον Δεκέμβριο κατάφερε να πάρει την πρωτοβουλία να εργαστεί όχι μόνο του εμπλεκόμενου στη χώρα, αλλά και με τι τοπικές αρχές, που είναι πολύ σημαντικό Όσοι ξέρετε την κατάσταση, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να δουλεύει κανείς σε διάφορα μέτωπα παράλληλα. Και αυτός εργάζεται, κάνει ένα πολυμέτωπο αγώνα, ξέρει να διαπραγματεύεται, θα πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Ε, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο δεν μπορεί να τα κάνει αυτά μόνη της. Χρειάζεται την υποστήριξη τη ε, Διεθνούς Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, αλλά και των ε, μελών του Συμβουλίου Ασφαλεία στη Νέα Υόρκη. Πιστεύω ότι όπως αναφέρατε και πολλοί από εσά, το θέμα της ε, ανθρωπιστικής κρίσης είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί σε μια κατακαιρματισμένη κατάσταση ασφαλείας αυτό που συμβαίνει πάντα είναι οι πολίτες της χώρας ε, πέφτουν θύματα και πληρώνουν αυτή το μεγαλύτερο τίμημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ε, κανένας νόμος του διεθνούς δικαίου δεν γίνεται σοβαρός και το να ε, προωθηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια είναι τεράστιο ε, πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά είμαστε μεγαλύτεροι ε, δωρητές. Ε, πέρα από την ΕΚΟ διάφορα εργαλεία έχουν αναθεωρηθεί ούτω ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των μεταναστών και των πολιτών της Λιβύης. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει η βοήθεια αυτή σε όλους, αλλά νομίζω ότι είμαστε ο πιο ενεργός φορέας ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την τρομερή ανθρωπιστική κρίση και ανάγκη. Ε, τώρα, για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν προσπαθούμε να προωθήσουμε μια πολιτική λύση, όταν βλέπουμε τι κινδύνους αντιμετωπίζει η Λιβύη, συνειδητοποιούμε ότι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, βλέποντας τις ε, διάφορες πολιτοφυλακές που δραστηριοποιούνται στη Λιβύη, το πώς ελέγχουν ε, τον πληθυσμό και τους αμάχους, το πώς ε, παραβιάζουν τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι σημαντικό να ζητάμε όχι να δοθεί προσοχή μόνο σε αυτό, αλλά να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Και δεν αμφιβάλλω ότι το μέγιστο αυτό μπορεί να γίνει αν υπάρξει πρόοδος ε, στις συζητήσεις για τη νέα κυβέρνηση και για το σχηματισμό της κυβέρνησης, πόσα μέλη θα έχει, όλα αυτά τα θέματα που είναι σημαντικά τώρα. Ε, δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα αλλά μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα έγινε για να δει τι ακριβώς ε, συμβαίνει επί τόπου. Θα πρέπει να καταρτήσουμε επίσης και ανθρώπους, ούτω ώστε ε, οι δημοσιογράφοι να αναφέρουν τις παραβιάσεις ε, των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα που αφορούν την διαδικασία αυτή μετάβαση σε μια ασφαλέστερη κατάσταση για λόγους έτσι, χρόνου δεν θα επεκταθώ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, χωρίς αφελείς πεπιθήσεις, όπως είπε και το Κοινοβούλιο, αλλά συνειδητοποιώντας ότι η πολιτική λύση και στη Λιβύη, Λιβύη όπως και αλλού, είναι η πιο αποτελεσματική. Δεν είναι μια ήπια προσέγγιση, είναι μια απόπειρα για να υπάρξει κάποια τάξη. Δεν πρόκειται ξαφνικά να γίνει Λιβύη Δανία, ας πούμε αλλά μια, ένα πρώτο βήμα για να βρει ξανά την σταθερότητα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να αντιμετωπίσει την απειλή του ISIS και άλλων εξτρεμιστών. Ευχαριστώ. Έχουμε λάβει 8 προτάσεις ψηφίσματος που έχουν πρόθεσμα κατατεθεί. Η συζήτηση έχει κλείσει.